Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να σας μιλήσω σήμερα το πρωί. Ε, εμείς πρόσφατα ε, δημοσιεύσαμε μια γνωμοδότηση που αφορά στις προϋποθέσεις του άρθρου 33.2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι πώς αυτά ε, εφαρμόζονται σε ενωσιακό πλαίσιο και πώς αντιμετωπίζεται η λειτουργία του ενωσιακού πλαισίου για να προάγει, να προστατεύει και να ελέγχει ε, την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση ε, επιμερίζει τις ε, προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33.2 της ε, Σύμβασης των Εθνών μέσα σε ενωσιακό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζει νομικής φύσεως θέματα, δηλαδή το ποιος πρέπει να εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ε, πώς πρέπει να γίνεται ο ορισμός και η προστασία, αλλά εξετάζονται και πρακτικά θέματα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνεται από το πλαίσιο ή μέσα στο πλαίσιο και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση είναι το αποτέλεσμα ενός αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προήλθε αρχικά από αυτήν την Επιτροπή. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που και εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις νομικές μας γνώσεις στη δουλειά του Κοινοβουλίου για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ελπίζουμε η γνωμοδότηση να στηρίξει τελικά τις ε, προετοιμασίες για την έκθεση που αφορά στην εφαρμογή του CPRD και της Επιτροπής του, ε, μια έκθεση που δημοσιεύτηκε πέρυσι. Ακούσαμε πολύ συχνά την σημασία της ε, σύμβασης όσον αφορά την ε, αναπηρία και θέματα ανισότητας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι πολίτες με ίσα δικαιώματα να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως ε, στην κοινωνία. Και αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι οι, τα κριτήρια που αναφέρονται στη σύμβαση θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προϋποθέτει πάλι την ε, ε, συμμετοχή πολλών φορέων, αλλά ο φορέας που παίζει ε, καθοριστικό ρόλο είναι αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή, την προστασία και τον έλεγχο των διατάξεων της Σύμβασης. Αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το τρέχον πλαίσιο, γιατί σας είπα και εμείς είμαστε μέλη αυτού του πλαισίου. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να εστιάσω την προσοχή μου σε τέσσερα παραδείγματα για το τι ακριβώς ε, σημαίνει το να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της ε, σύμβασης, κυρίως αναφορά την πλήρη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν όσον αφορά στην νομική βάση του πλαισίου πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια, τη νομική βεβαιότητα και την προβλεψιμότητα. Και εμείς πιστεύουμε ότι ε, ένας ε, νομικά, ε, μια δέσμευση νομική, αυτό μπορεί να αποτελεί τη νομική βάση και να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτά μπορούν να γίνουν με διαφορετικές μορφές. Μία λύση είναι η αναθεώρηση του υπάρχοντος κώδικα συμπεριφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία και η εκπροσώπηση της Επιτροπής μας. Ένα άλλο θέμα μια άλλη εναλλακτική λύση είναι μια διοργανική συμφωνία. Και τρίτη λύση θα μπορούσε να είναι λήψη απόφασης που θα διευκρινίζει ε, συγκεκριμένα στοιχεία των βασικών ε, λειτουργιών του κώδικα. Ένα θέμα λοιπόν που μπορεί να διευκρινίσει μια τέτοια νομική πράξη είναι η σύνθεση και η διαμόρφωση του πλαισίου. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή αποτελείται από τέσσερις οργανισμούς. Ένας εξ αυτών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά έχουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Οργανισμό για Θεμελιώδη Δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για ε, άτομα με αναπηρία και ο Ευρωπαϊκός Φορέας και ο Διαμεσολαβητής ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητοι μηχανισμοί που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο όπως ακριβώς προβλέπει η συνθήκη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης ε, και αυτό εκφράζει τις ε, αρχές των Παρισίων που αφορούν στη σύσταση και τη λειτουργία θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για τον πλουραλισμό και για τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων και εμπλεκομένων στη διαδικασία ελέγχου. Όσον αφορά στην πολυμορφία, για να εκφράζεται αυτή στην κοινωνία και να αφορά και στους φορείς που, που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του ε, πλαισίου. Για να υπάρχει αυτή η πολυμορφία θα έπρεπε να συσταθεί μια συμβουλευτική επιτροπή και με αυτήν ε, το πλαίσιο θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με διάφορους φορείς. Ένα τρίτο ε, κομβικό στοιχείο της γνωμοδότησης αφορά στα καθήκοντα του ενωσιακού πλαισίου που μπορούν να κατατμηθούν σε τρεις βασικούς τομείς. Ένας εξ αυτών είναι η προαγωγή, η προστασία και ο έλεγχος και ε, η γνωμοδότησή μας κατατείνει στο ότι τα βασικά στοιχεία αυτών των τριών τομέων μπορούν επίσης να διευκρινιστούν τουλάχιστον όσον αφορά τη νομική τους βάση. Όσον αφορά στην προαγωγή Υπάρχουν πάρα πολλές ε, δραστηριότητες οι οποίες ε, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιπτώσεις από διάφορα μέλη του πλαισίου. Εδώ περιλαμβάνεται η δημιουργία δυνατοτήτων, ε, ο εξονυχιστικός έλεγχος της κείμενη νομοθεσίας, κατά πόσον αυτή είναι συμβατή και επίσης και το κατά πόσον εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σύμβαση. Δεύτερον, όσον αφορά στην προστασία, εκεί ε, μπορεί να υπάρξει έρευνα και έλεγχος ενστάσεων ή δυνατότητα να γίνονται έρευνες και να συγκεντρώνονται δεδομένα, όπως επίσης και να υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή να διεξάγονται έρευνες και μετά από την πρωτοβουλία του ίδιου του πλαισίου, κατόπιν να μπορούν να δημοσιεύονται ε, εκθέσεις που να αφορούν στην εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία, του CTP, αντί όπως αναφέραμε προηγουμένως. Η ανάλυση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, παράλληλα με δείκτες ε, και συγκριτικά στοιχεία για να μπορεί κανείς να αξιολογήσει την εφαρμογή της ε, σύμβασης. Να υπάρχουν και μελέτες και σε τομείς όπου υπάρχει στασιμότητα ή ακόμα και οπισθοχώρηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει σχέση με τον έλεγχο είναι η ενεργός συμμετοχή του πλαισίου στη διαδικασία αναθεώρησης από την Επιτροπή της Σύμβασης. Και αυτό περιλαμβάνει και την υποβολή εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Ένα τέταρτο θεμελιώδες στοιχείο ε, που έχει ε, που έχει άμεση σχέση με τα καθήκοντα είναι το εξή. Το να εξετάσει κανεί ε, το κατά πόσον υπάρχουν επιπρόσθετοι πόροι έτσι ώστε το πλαίσιο να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του η ανάγκη για τέτοιους επιπρόσθετους πόρους ε, επισημάνθηκε κυρίως από την Επιτροπή της Σύμβασης ε, στις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση λοιπόν που μία νομική πράξη αναφέρει με σαφήνεια ποια είναι αυτά τα καθήκοντα, η δική μας άποψη είναι ότι είναι σημαντικό να ελέγξουμε κατά πόσον πρόκειται για νέα και επιπρόσθετα καθήκοντα για τα μέλη ε, του πλαισίου, ε, γιατί αν πρόκειται κάτι τέτοιο, αυτό προσαφώς και προϋποθέτει επιπρόσθετους πόρους. Τι είναι λοιπόν, τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Η ε, σημασία αυτής της γνωμοδότησης βρίσκεται στις καταληκτικές παρατηρήσεις ε, της Επιτροπής της Σύμβασης σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για παρατηρήσεις που έχουν σχέση με το πλαίσιο και ε, με την εφαρμογή του πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης και με το κατά πόσον γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος, ε, όπως και σε όλες τις ε, καταληκτικές Και εδώ βλέπουμε ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Εμείς ελπίζουμε η γνωμοδότηση αυτή να ταιριάξει στην συνέχιση εφαρμογής της σύστασης τη σύμβαση με συγχωρείτε, μάλλον των συστάσεων, κυρίως το άρθρο 33. Ε, πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβατή με τη σύμβαση και κατά πόσον έχει ένα ελεγκτικό μηχανισμό, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το να υπάρχει ένα ουσιαστικό πλαίσιο που θα προάγει, θα στηρίζει, θα προστατεύει και θα ελέγχει την εφαρμογή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει, από αυτό συνάγεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει στα σοβαρά τις υποχρώσεις της. Επειδή η σύμβαση είναι η πρώτη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπρόσθετα από τα κράτη-μέλη, είναι δηλαδή συμβαλόμενο μέρος, είναι σημαντικό να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει να πράξει τα δέοντα για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο της σύμβασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Μάρκ Πλούρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις ε, και δικές μου αλλά και του κυρίου Άνταμ Κόσα που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στην διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών της σύμβασης στη Νέα Υόρκη. Ομολογώ ότι μάλλον είμαστε απογοητευμένοι από την ε, έκθεση που ετοίμασε ο Οργανισμός Θεμελών Δικαιωμάτων με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε πιο διαφανή ε, παρουσίαση των θεμάτων. Έχουμε πολλές επιφυλάξεις για την έκθεση αυτή θεωρώ ότι δεν έχουμε στην έκθεση αυτή εμβριθεί ανάλυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, ε, παραλείπεται τελείως το γεγονός ότι ε, συμμετέχουν όχι μόνο η Επιτροπή Αναφορών, αλλά και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η Επιτροπή ε, Απασχόλησης εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό, και, εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, στο σημείο 26 με 28, δυστυχώς δεν αναφέρεται σωστό ρόλο ρόλος του Ευρωπαϊκού και αυτό μας ε, ευνηδιάζει και μας απογοητεύει. Επίσης, ε, έχουμε την εσωτερική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ότι δραστηριότητες γίνονται σε κάθε συγκεκριμένο τομέα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο ΦΡΑ, με αυθαίρετο τρόπο διαπιστώνει ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός ε, των ε, αρμοδίων τέτοιων σωμάτων. Θα έπρεπε η έκθεση να επικεντρώνεται κυρίως στο ρόλο του οργανισμού των θεμελιών δικαιωμάτων, του ίδιου του ΦΡΑ. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η ε, παρουσίαση που γίνεται από την άποψη αυτή. Και ο Άνταμ Κόσα, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ επικριτικά κρίνουμε αυτή την έκθεση του, του οργανισμού ΦΡΑ. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, λοιπόν Πρόεδρος, και θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μιλκεβιζιούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Θερμιδών Δικαιωμάτων για την παρακολούθηση του CTRPD στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, διαμόρφωση και τη δομή του Ευρωπαϊκού Σχετικού Πλαισίου. Και θα ήθελα αυτή τη φορά να υποστηρίξω τον συνάδελφο Πλουρά. Να πω δε ότι η γνωμοδότηση του ΦΡΑ για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ανησυχεί σε κάποιο βαθμό και δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να την υποστηρίξω. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει ότι η Επιτροπή ή το Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσουν το ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση του πλαισίου. Το έχουμε αυτό ήδη αναφέρει σε σχετικό ψήφισμα στις 28 Μαΐου του 2015. Είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Αυτοπλασίου. Ως εκ τούτου έχει δικαίωμα να λαμβάνει τις του αποφάσεις για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και για το ποιες ε, επιτροπές θα πρέπει να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του CT, του PRD η Επιτροπή Αναφορών. Έχουμε υποφανθεί ότι δεν επαρκεί και ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και Δικαιωμάτων του Πολίτη θα πρέπει να εμπλακούν. Ε, πιστεύω ότι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να αποφασίζουμε σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθηση. Αυτό ήθελα να πω στην παρούσα φάση, αλλά εκ νέου θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι ανεξάρτητη δομή και από μόνο του αποφασίζει ποιε επιτροπέ θα το εκπροσωπήσουν. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακολούθηση της σύμβασης CBRD. Σα ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στην κυρία Κούνεβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Στίκινγκς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για την δουλειά που έκανε ο οργανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ένας οργανισμός που αρκετά συχνά δημοσιεύει πολύ καλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα τα οποία απορώ γιατί δεν λαμβάνομαι περισσότερα υπόψη. Θα ήθελα με την σειρά μου να μοιραστώ και τις δικές μου σκέψεις με αφορμή την γνωμοδότηση. Το κείμενο που μας παρουσιάστηκε σήμερα λέει δυστυχώς το αυτονόητο. Γιατί λέω δυστυχώς, γιατί με λύπη διαπιστώνω και μέσα από την δουλειά που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την καθημερινή ζωή, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Κομισιόν και το Συμβούλιο κοφεύουν όταν καλούνται να εφαρμόσουν πραγματικά κοινωνικές πολιτικές. Δεν γίνεται να βρισκόμαστε μπροστά στο τόσο σημαντικό γεγονός της κυρώσης μιας τόσο σπουδαίας διεθνούς συμβάσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία οντότητα και την ίδια στιγμή να επισημαίνει η Κομισιόν πώς τα περισσότερα μέτρα που χρειάζονται για την εφαρμογή της είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αφού το ανακαλύπτει να μην κάνει καμία κίνηση για να δεσμεύσει τα κράτη-μέλη της ώστε να κινηθούν στην κατεύθυνση να λάβουν τα απαραίτητα αυτά μέτρα. Να σας πω όμως πως φοβάμαι ότι η Κομισιόν δεν θα προχωρήσει σε μια επί της ουσίας ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας. Και δεν μπορώ παρά να πω πως η στάση της είναι τουλάχιστον υποκριτική. Το λέω αυτό γιατί όταν πρόκειται για τις δημοσιονομικές πολιτικές η Κομισιόν παρουσιάζεται πάντα άκαμπτη. Τώρα που πρόκειται για θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων ανακαλύπτει ένα σωρό διοικητικά και νομικά καλύματα. Αυτά που μας λέει στην ουσία είναι ότι δεν μπορεί να επιβάλλει κοινέ πολιτικές. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος η σύμβαση του ΟΗΕ να εφαρμοστεί επιλεκτικά και να γίνει προνόμιο μόνο των πλούσιων κρατών της Ένωσης. Και όπως ακούσαμε ήδη, την ανάγκη για νομικά δεσμευτική πράξη από πλευρά της Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση, την επισημαίνει στην γνωμοδότηση του και ο οργανισμό για τα τεμιλιώδη δικαιώματα. Και αυτό όχι μόνο για να δεσμεύσει τα κράτη-μέλη για να αναλάβουν την απαραίτητη δράση, αλλά και να καθορίσει σε σαφήνεια, με σαφήνεια μια σειρά από θέματα που θολά στο πλαίσιο της λειτουργίας τους υπάρχοντος ευρωπαϊκού πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης, όπως το ποιος έχει την ιδιότητα μέλους και τι είδους μέλους, πώς θα εμπλακούν περισσότερο οι οργανώσεις ΑΜΕΑ και των σχετικών με τη Σύμβαση Φορέων. Νομίζω είναι σαφές πως και από την πλευρά μας έχοντας και την γνωμοδότηση αυτή στη φαρέτρα, μας πρέπει να πιέσουμε ώστε να αναλάβει επιτέλους την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία η Κομισιόν. Επίσης, την νομοδότηση του οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχουν ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επικοινωνίας μέσα σε κάθε κυβέρνηση, αλλά και ανεξάρτητοι μηχανισμοί, ώστε να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο οριζόντια και κάθετα όσα προβλέπεται στη σύμβαση. Αναρωτέμαι όμως πώς μπορεί να γίνει επί της ουσίας εφαρμογή σε χώρες όπως η Ελλάδα, στις οποίες ο διοικητικός μηχανισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες και πολλά από τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ έχουν θυσιαστεί στο βωμό της λιτότητας και είναι μια λιτότητα δεσμοποιημένη. Επιβάλλεται δηλαδή από τους σκληρούς κανόνες για τα δημοσιονομικά. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας είμαστε ειλικρινές. Η σύμβαση ΑΜΕΑ και καμία άλλη σύμβαση και κείμενο που προωθεί και προσπαθεί, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρόκειται στην ουσία ποτέ να εφαρμοστεί αν πρώτα δεν σταματήσουμε τις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στις οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω πολύ σύντομα για ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει αναφερθεί και στην γνωμοδότηση την, κατασκευή του σελίδα που τα αφορά τη λειτουργία και τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού πλαίσιο Εφαρμογή. Αναφέρεται στην γνωμοδότηση πω η ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά με σχετικές την εφαρμογή της Συμβάσης ΑΜΕΑ, πληροφορίες και γεγονότα. Η σελίδα αυτή θεωρώ θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο ιστοσελίδας και να είναι προσβάσιμη και αναγνωρίσιμη από ΑΜΕΑ, όχι μόνο όπως άλλες ε, σελίδες οργάνων και οργανών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για να τις διαβάσει π.χ. ένα άτομο με μειωμένη όραση πρέπει να έχει εγκαταστήσει ειδική εφαρμογή στο κινητό του. Από κατασκευή της ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης και σε κάθε δυνατή μορφή που εξυπηρετεί τις ανάγκες αμαία. Κλείνοντας, το είχε πει και θα το ξαναπώ. Δίνουμε εξετάσεις ως Ένωση. Η εφαρμογή του σπουδαίου κείμενου της Συμβάσης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την ίδια την Ένωση. Σε περίπτωση μη κατολικής και ομοιόμορφης εφαρμογής της, στις χώρες της Ευρώπης θα έχουμε θυσιάσει τα δικαιώματα στα άτομα των ισοσκελετισμένων και πλεονασματικών προϋπολογισμών. Θα έχουμε μια οικονομία που δουλεύει εις βάρος των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους. Αν όμως επιτύχουμε την πραγματική εφαρμογή της συμβάσης, θα έχουμε κάνει ένα σοβαρό βήμα για να τεμιλιώσουμε μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΧΟΜ ίσως και μήπως θα θέλετε να απαντήσετε και να σχολιάσετε αυτή την έντονη κριτική. Είναι εδώ οι συνάδελφοι και θέλουν να πάρουν το λόγο για να απαντήσουν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους βουλευτές για τη γνώμη και την άποψη που μας παρουσίασαν. Την σημειώσαμε. Δυστυχώ οι εμπειρογνώμονε μα για το θέμα αυτό δεν μπορεί να παρευρεθούν εδώ σήμερα, γιατί όπω αναφέρθηκε και προηγουμένω, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την διάσκεψη των ημερών. Ω εκ τούτου, θα διαβασφαλίσουμε ότι όλα σα τα σχόλια θα, σας, ε, θα τους διαβιβαστούν προκειμένου και να ληφθούν υπόψη για τις μελλοντικές τους εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στίκινγκς, ε, έχετε κάτι να προσθέσετε? Σας ευχαριστώ πολύ, να σας ευχαριστήσω και για τα σχόλια που κάνατε. Ξεκινώντας ε, με το θέμα που, έστει, που έθεσε η κυρία Κινέβης για το, την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα για το πλαίσιο έχει ήδη δημιουργηθεί και διατίθεται εν μέρη στο, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ΒΡΑ, αλλά προφανώς αποτελεί ένα κομμάτι ενός συνόλου σε ό,τι αφορά την προσπαθμότητα τώρα της ιστοσελίδας. Υπάρχει και η νοηματική γλώσσα και παροχή easy της, ε, των πληροφοριών και στο σύνολο της ε, η ιστοσελίδα του ΦΡΑ προσπαθεί να πληρεί τα, τους όρους και τις συνθήκες ε, της CTRPD 2.0. Προφανώς, πάντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που θα γίνουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τα άλλα σημεία που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο. Νομίζω ότι η ιδέα της νομικής βάσης είναι να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια στη σύνθεση της συμμετοχής ε, στις δραστηριότητες του πλαισίου και ούτω καθεξής. Ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε, δεδομένων και των αλλαγών ε, στη σύνθεση του πλαισίου που έγιναν από τότε που αρχικά έγινε αποδεκτό το αρχικό σημείωμα στο 2012 από το Συμβούλιο με τη συμπερίληψη και άλλων επιτροπών. Λοιπόν, Υπάρχει λοιπόν η προοπτική να υπάρχει και ένα ανανεωμένο νομικό έγγραφο που θα αποτυπώνει αυτές τις ενημερώσεις. Αυτό δεν θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου, αλλά θα δώσει σε αυτό το σημαντικό σώμα, το οποίο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, και την νομική βεβαιότητα και τη βιωσιμότητα που πραγματικά χρειάζονται για να υποστηρίξουν το έργο της προστασίας και της παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, κανονικά δεν είμαστε ούτε τόσο αμήλικτοι, ούτε τόσο δρεμοί στην κριτική μας ε, εδώ από πλευρά της Επιτροπής μας όσο είμαστε για το συγκεκριμένο θέμα. Προσβλέπουμε ωστόσο στις μεραδικέ μας επικοινωνίε και συζητήσει για το θέμα αυτό. Και μετά από αυτά, να ευχαριστήσουμε όλους ε, τους συμμετέχοντες για το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 16 στην ημερήσια διάταξη για την ίδρυση του, προγράμματος υποστηρίξης συντηρητικών μεταρρυθμίσεων για την ε, περίοδο 2017-2020. Αν είναι εδώ η κυρία Μακάρθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πάρει το λόγο. Αν θα θέλετε να μας κάνετε μια εισαγωγή στις εργασίες αυτές για τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Κανείς όμως δεν είναι εδώ, σχολιάζει ο Πρόεδρος, για να πάρει το λόγο. Okay, then Μάλιστα, να δώσουμε τον ε, λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Τσάμπα Σόγκουρου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου που είδα τις τελευταίες συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ότι υπάρχει μεγάλη ε, έμφαση στα θέματα τα κοινωνικά και στα θέματα της ενεργείας. Και πιστεύω ότι πέρα από την, ε, τα δημοσιονομικά και τη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και θέσεων Απασχόληση χρειαζόμαστε διαφορετικέ μεταρρυθμίσει και στον τομέα των κοινωνικών. Και όπω είπε και η κυρία Τάισεν αυτή την εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, μόνο αν ληφθούν υπόψη κοινωνικέ διαστάσει σε όλου του τομεί τη πολιτική θα καταφέρουμε πραγματικά να πετύχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Η ανάγκη για τι μεταρρυθμίσει λοιπόν είναι πιο επιτακτική παραποτέ σήμερα. Η οικονομική ανάπτυξη ανησυχητική και τα οικονομικά μεγέθη και η οικονομική αυτή η κρίση στραβλώνει όλους πιο πολλούς ε, τομείς της ζωής σήμερα. Προκειμένου λοιπόν να, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη μεταρρύθμιση στο θέμα της ε, εκπαίδευσης και για την νομοθεσία για την αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν η δημιουργία ενός μόνιμου προγράμματος υποστήριξης ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ξεχωριστό προϋπολογισμό θα είναι τόσο σημαντικός και το χαμηλός βαθμός ε, εφαρμογής της νομοθεσίας της ERS από διάφορα κράτη-μέλη αποτελούν εμπόδιο για τις επενδύσεις και για την δημιουργία ενό φιλικού περιβάλλοντος προς τις ε, θέσεις εργασίας. Φυσικά, δεδομένου και των ε, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κρατών μελών, κάποιες χώρε θα επωφελούνταν πιο πολύ από την υποστήριξη αυτή από παρά άλλε. όπως η Ρουμανία, η δική μου χώρα, όπου περιορίζεται η πολυπλοκότητα τη διοικητικών διαδικασιών. Αν υπήρχε λοιπόν τέτοια υποστήριξη εκ των προτέρων για τη χώρα μας, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε τόσο χαμηλό βαθμό φυτικότητα των πόρων σε ύψους 70% για την περίοδο την τελευταία. Και θα είχαμε χάσει τόσο πολύτιμο χρόνο. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την προγραμματική περίοδο και σε ό,τι αφορά τι θεσοδικές μεταρρυθμίσει δεδομένων και συμπεριλαμβανομένων των ε, α, συμφωνιών εταιρετικών σχέσεων. Και νομίζω ότι εν μέρη ε, Έλεψε η στρατηγική σε διάφορους σημαντικούς και ουσιώδες τομείς, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Κάποια ερωτήματα τώρα. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει φυσικά κανεί για να ακούσει τα ερωτήματα αυτά. Καταρχά, ε, η πρόταση είναι εγγενώ περίπλοκη. Καλύπτει και το EFS, το EFSI, του EFSI και τι μακροοικονομικέ προσεγγίσεις και διαστάσει εκ Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την περιπλοκότητα και πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε με την χρηματοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή. Και των δεύτερον, πώ θα εξασφαλίσετε ότι η τυπική αυτοδιοίκηση θα ωφεληθεί επίση από την υποστήριξη αυτή και όχι μόνο η κεντρική κυβέρνηση. Και τρίτον, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη έχουν τεχνική αρρωγή από τα εθνικά ταμεία προ υποστήριξή του για τη χρηματοδότηση τέτοιων ενεργειών υποστήριξη στην πράξη, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε περιπτώσεις διπλής χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μα τι γίνεται. Έχουμε όχι Brexit, αλλά exit στην Επιτροπή μας. Δεν έχουμε γεμάτους καταλόγους ε, ομιλητών ως συνήθως. Η κυρία Χάρκιν, μήπως εκπροσωπεί την ομάδα τη. Αλλά, Σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, ε, για να είμαι ειλικρινής, ε, κυρία Πρόεδρε, ε, θέλω να σα πω ότι θα ήθελα να είναι εδώ η Κομισιόν, γιατί θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσει. Πάντω, εγώ ε, δεν το ήξερα το θέμα, το διάβασα πάρα πολύ γρήγορα και από ό,τι φαίνεται θα γίνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, τα κράτη-μέλη ε, μπορούν και πρέπει να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους, τι διοικητικές κυρίω. και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σε κάποια κρατημέλη τα, κρατη, τα κρατημέλη θα αποφεληθούν από ορισμένους τομείς περισσότερο. Θα υπάρχουν πάντως ευκαιρίες για όλα τα κρατημέλη για να αποφεληθούν από αυτές τις προτάσεις. Και νομίζω θα υπάρξουν και οικονομίες κλίμακας. Σε αυτή την Επιτροπή μιλάμε συχνά για τις βέλτιστες πρακτικές, πώς μπορεί κανείς να επωφεληθεί από αυτές ε, αυτός είναι ένας τρόπος για να πάρει μια τυπική μορφή το θέμα. Ε, πράγματι, θα πρέπει να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα και επειδή αναφέρατε το θέμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία, μετά από ακριβώς μια εβδομάδα οι Βρετανοί θα αποφασίσουν. Με εν πάση περιπτώσει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα και πραγματικά ελπίζω να αποφασίσουν οι Βρετανοί να παραμείνουμε, νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα μάθημα για όλους μας ότι αν γενικά οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ένα όραμα για την κοινωνική Ευρώπη, το οποίο όμως και να εφαρμόζεται, τότε η αφοσίωση και η πρόσδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια τόσο ισχυρή. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι το εξή. Μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι πάντα όταν ακούω αυτόν τον όρο ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί θέλω να ξέρω ακριβώς για το τι πράγμα μιλάμε. Γιατί μπορεί κανείς να μιλήσει σε δύο ε, διαφορετικούς ανθρώπους και να έχουν ε, διαφορετική πολιτική προσέγγιση και αυτοί έχουν και δύο ε, διαφορετικές απαντήσεις για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μιλάμε όμως όλοι για το ίδιο πράγμα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω πολλές ειδικέ γνώσεις επί του θέματος, αλλά όπως σας είπα είχα ελπίσει να ακούσω κάποια πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πάντως θέλω να συμβάλλω στη συζήτηση και προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή τον κύριο Σόγκα. Ο κύριος Περίνσκι αντικαθιστά το συνάδελφό του. Δεν ξέρω, μήπως να ακούσουμε ε, καλύτερα πρώτα την Κομισιόν και μετά να επανέλθετε, γιατί Έχουμε την κυρία Μαρία Μακάτι εδώ μαζί μας. Ένα λεπτό μπορείτε να έχετε για να καθίσετε και μετά με πολύ μεγάλη χαρά να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Όταν ετοιμαστείτε πέστε μας για να ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα των... Ε, στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πρόταση μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο για την ακρίβεια πέρυσι, υιοθέτησε μία πρόταση για τη στήριξη προγραμμάτων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως τμήμα του, της δέσμης μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για ποιο λόγο υποβάλαμε αυτή την πρόταση. Στόχος του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι να διαφυρώσει κάποια κανονιστικά κενά που παρατηρήθηκαν στα κράτη-μέλη ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μας ενδιαφέρουν είναι κυρίως αυτές που γίνονται στο πλαίσιο των ειδικών συστάσεων αναχώρα. Αλλά δεν περιορίζονται στις ειδικές συστάσεις αναχώρα οι διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις. Η στήριξη, η τεχνική συνδρομή που προσφέρουμε στα κράτη-μέλη προβλέπει τεχνική συνδρομή και στα πλαίσια της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Τους κύκλους παραβίασης και άλλες κυβερνητικές διαδικασίες όπως είναι η Ενεργειακή, η Ενεργειακή Ένωση και η Ένωση Κεφαλαγορών. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο στις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Τώρα, το είδος της αρρωγής που προβλέπουμε, της τεχνικής συνδρομής που προβλέπουμε, είναι συγκεκριμένη συνδρομή προς τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ανάγκες ε, του συγκεκριμένου κράτους κυρίως για να συμπληρωθεί η διοικητική ικανότητα του κράτους επιτόπου. Η εντολή που έχουμε περιλαμβάνει όχι μόνο τέτοιου είδους συνδρομή, για την εφαρμογή δηλαδή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά ταυτόχρονα και συνδρομή, στήριξη, προκειμένου να αξιοποιηθούν ε, αποτελεσματικά και στο έπακρο τα διαρθρωτικά κονδύλια. Η διάρκεια της πρότασης είναι τετραετής και καλύπτει την περίοδο 2017-2020. Το προτινόμενο ποσό που προβλέπετε είναι 142,8 εκατομμύρια ευρώ. Περνάμε τώρα στους στόχους της του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο γενικός στόχος που αναφέρεται στην πρόταση είναι η ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να προετοιμάσουν ε, μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη μέσω της ε, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Αυτός είναι ο γενικός στόχος. Περνάμε τώρα στους ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν ε, την στήριξη των εθνικών αρχών των κρατών μελών με πολλούς και διάφορους τρόπους. Στηρίζουμε τις εθνικές αρχές μέσω κάποιας τεχνικής συνδρομής για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν τις μεταρρυθμίσεις ανάλογα με τις προτεραιότητές τους. Επίσης, προβλέπεται συνδρομή για να ενισχυθεί η ικανότητα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Επίσης, ε, τους στηρίζουμε στον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και μεθοδολογιών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό, γιατί η ιδέα των βέλτιστων πρακτικών ήδη υπάρχει, αλλά στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί από τα κράτη-μέλη και Δηλαδή να μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ευέλτιστες πρακτικές χωρών που έχουν παρόμοιες συνθήκες. Και τέλος, ε, τελευταίος ειδικό στόχος είναι η ενίσχυση της διαχείρισης ε, του ανθρώπινου δυναμικού, των ανθρώπινων πόρων. Ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι τι είδου στήριξη προσφέρεται σε τι συνίσταται αυτή η στήριξη, η τεχνική συνδρομή που προβλέπεται μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η στήριξη έγκυται στην παροχή συνδρομής ε, στα κράτη-μέλη, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, είτε άμεσα μέσω των εμπειρογνωμόνων μας, γιατί έχουμε εμπειρογνώμονες για διάφορους τομείς. Επίσης έχουμε εμπειρογνωμο... εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορούμε να την κινητοποιήσουμε και να στείλουμε στα κράτη-μέλη, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αποστολές εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη. Τέτοιου αποστολές χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των προβλημάτων και για τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη ε, της ε, ακολουθητέας καλύτερης και πιο κατάλληλης μεθόδου. Αν τα κράτη-μέλη ήδη έχουν εκπονήσει την θεωρητικά τη μεταρρυθμίσή του, αλλά δεν έχουν εφαρμόσει, μπορούμε να παράσχουμε τεχνογνωσία οργανώνοντα σεμινάρια για να συζητήσουμε τον κατάλληλο τρόπο για την εφαρμογή των ελλημένων μεταρρυθμίσεων. Επίση, στέλνουμε πολλέ φορέ και εμπειρογνώμονες στη διοίκηση των κρατών μελών. Για παράδειγμα, μπορούμε πυρογνώμονε για συγκεκριμένο κλάδο να του στέλνουμε στα Υπουργεία ή σε άλλα τμήματα τη Δημόσια Διοίκηση για να βοηθήσουν σε συγκεκριμένα προγράμματα, στην ενέργεια, στη φορολογία, και ούτω καθεξής. Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε άμεσε επαφές με διεθνή Ινστιτούτα και οργανώσεις για να προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη και μέσω ε, δημοσίων συμβάσεων προσλαμβάνουμε εμπειρογνώμονες προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα, το εύρος της στήριξης, το πεδίο εφαρμογής. Είναι αρκετά ευρύ αυτό το πεδίο. Καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό τομέων. Απαριθμούνται εδώ στη διαφάνεια και περιλαμβάνουν τη φορολογία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ε, διαχείριση του φορολογικού εισοδήματος, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της απάτης, της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίση στο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, εμπόριο, ξένες ε, εμπορικές επενδύσεις, αηφόρος ανάπτυξη, Βρείτε το φάσμα λοιπόν της στήριξης και περιλάβαμε και κάποια συνδρομή στα πλαίσια των πολιτικών αγοράς εργασίας, κοινωνική συμπερίληψη, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια, γεωργικές πολιτικές. Ένα από τα νέα στοιχεία προβλέπει στήριξη και στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πώς ενεργοποιείται τώρα αυτή η στήριξη του προγράμματος το πρόγραμμα ενεργοποιείται με απλή αίτηση του κράτους μέλους. Δεν ε, υπάρχει καμία είδους επιβολή για την υποχρεωτική αποδοχή της στήριξης αυτής. Το κράτος μέλος ή και ο θελός υποβάλλει το αίτημα για παροχή στήριξης. Πρέπει να κάνει δηλαδή το κράτος μέλος το πρώτο βήμα και να ζητήσει αυτή τη στήριξη. Βέβαια δίνουμε κάποιες καθευθυντήριες γραμμές για το είδος του αιτήματο που θα ήταν παραδεκτό ή ευκταίο από τα κράτη-μέλη. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις ε, που ενεργοποιούν αυτό το αίτημα για την παροχή τεχνικής συνδρομής. Υπάρχουν τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, τα προγράμματα αυτά από κράτη-μέλη που έχουν μνημόνιο. Πρόκειται για μια συνέχιση της μεθοδολογίας που είχαμε στο παρελθόν με ε, τη Task Force που στείλαμε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εκεί είχαμε άμεση παροχή τεχνική συνδρομή στα δύο κράτη για να ε, εφαρμόσουν καλύτερα τα προγράμματα οικονομική προσαρμογή. Βέβαια τώρα επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα και σε όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια τη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Όπως είπα, τα κράτη-μέλη που έχουν ειδικέ στάσει σε ένα χώρα πολύ συχνά ζητούν τεχνική συνδρομή στον τομέα αυτό άλλη το του ενωσιακού δικαίου. Είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών, η Ενεργειακή Ένωση. Οπότε αιτήματα των χωρών στα πλαίσια αυτών των τομέων είναι παραδεκτές και θα ενεργοποιήσουν την τεχνική συνδρομή. Ένας άλλος παράγων είναι οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινούν τα κράτη-μέλη με δική τους πρωτοβουλία. Και αυτό θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν το πρόγραμμα στήριξης για την παροχή τεχνικής συνδρομής. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Από τη στιγμή που λάβουμε το αίτημα από το κράτος μέλος για την παροχή τεχνικής συνδρομής, το αναλύουμε υπό το φως των κριτηρίων που σας ανέφερα. Και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της ανάλυσης και της επεξεργασίας ενός αιτήματο είναι ο επίγον χαρακτήρας του προβλήματος. Μπορεί ένα κράτος να έχει μια προθεσμία για να εφαρμόσει συγκεκριμένη διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτή η χρονική πίεση θεωρείται όρος απαραίτητος, ο επίγον χαρακτήρας. Επίσης, η πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα κράτος και πρέπει να αντιμετωπίσει μια μακροχρόνια περίοδο, γιατί οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι και χρονοβόρε. Γίνεται μια ανάλυση λοιπόν του Εύρου και του βάθους του προβλήματος. Ένα κράτος, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί τεχνική συνδρομή σε συγκεκριμένο κλάδο, την αηφόρο ανάπτυξη, για παράδειγμα, την αηφόρο ενέργεια. Και επίση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στου κοινωνικο οικονομικού δείκτες, και τη γενική διοικητική ικανότητα του κράτους μέλους. Όταν ένα κράτος μέλος ζητά ιδιαίτερο είδος τεχνικής συνδρομής, εμείς εξετάζουμε κυρίως την ε, ε, ικανότητα, τη διοικητική ικανότητα που έχει ένα κράτος να απορροφήσει αυτή την τεχνική συνδρομή, γιατί δεν έχει νόημα να επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη με υπερβολική τεχνική συνδρομή, αν η ικανότητά τους να την απορροφήσουν είναι περιορισμένη. Περάμε τώρα στον προϋπολογισμό, το οικονομικό σκέλος του προγράμματος στήριξης διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Όπως είπα και προηγουμένως, θέλουμε να υπάρξει ένα εκτενές τέτοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης και προτείνουμε λοιπόν μέχρι 240 ε, εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν, αυτός ο φάκελος θα καλύψει όλη την τετραετή περίοδο και χρηματοδοτείται από την ε, εκ νέου χρήση του FS και του ERFD e, e και σε σε ό,τι αφορά τους νέους πόρους από πλευράς των κρατών, ε, μάλλον δεν πρόκειται για, ε, για καινούργιους πόρους, μιλάμε για εκ νέου χρήση μη ε, μη ε, χρησιμοποιημένων πόρων. Πρόκειται για ε, προϋπολογισμό της κεντρικής τεχνικής αρρωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ιδιαίτερος, οι πόροι τους οποίους έχουμε υπόψη μας είναι οι εξή από τον κεφάλαιο, την επικεφαλίδα 1β, 112,2 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό θα προέλθει από το ESF, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής. Από την επικεφαλίδα, ε, από τον τομέα 2, 30,6 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την ανάπτυξη της Υπέθρου. Πέρα από τους πόρους λοιπόν που ήδη διατίθενται, υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να επιστρέψουν από μόνα τους ε, αμα, πόρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο SRSS, για να ε, δοθούν από αυτά. Υπό το άρθρο υπαριθμών 35 του κανονισμού. Τα κράτη-μέλη προβλέπεται ότι μπορούν εφόσον του επιθυμούν, να μεταφέρουν και, να επιστρέψουν χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΣΡΕΣ για να χρησιμοποιηθούν εξ ονόματός τους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό ήδη εφαρμόζεται για χώρες που είναι σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Οι αρχές της Ελλάδας, για παράδειγμα, επέστρεψαν 15 εκατομμύρια στην Task Force για την Ελλάδα όπως ε, ονομαζόταν τότε, για να χρησιμοποιηθούν εξ ονόματος της Ελλάδος για τεχνική αρρωγή. Φέτος, δε, οι ελληνικές χαρχές μετέφεραν και επέστρεψαν 30 εκατομμύρια στο SRSS ε, για να ε, δοθεί τεχνική αρρωγή. Η διαφορά είναι ότι η δυνατότητα αυτή επιστροφής χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχει ε, δοθεί, επεκταθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς θα εφαρμοστεί λοιπόν το SRSP. Το SRSP θα ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Κανονισμό. Για το ρόλο λοιπόν του SRSP Έχουμε καταρτήσει πολυετή προγράμματα εργασία, τα οποία και θα αναλύουν τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την τεχνική αρρωγή, η οποία θα χορηγηθεί και θα περιλαμβάνουν και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της τεχνικής αρρωγής, θα ορίσουν τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στους εκάστοτε τομείς της πολιτικής και πέρα από τα πολυετή προγράμματα εργασίας καταρτίζονται και θα λαμβάνονται και αιτήσει αποφάσεις. Το συνολικό ποσό είναι 142,8 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Αλλά για κάθε χρόνο θα προβλέπετε ένα ποσό για την ε, παροχή τεχνικής αρρωγής για το συγκεκριμένο έτος. Το ποσό δε αυτό θα βασίζεται στα αιτήματα τα οποία θα λαμβάνουμε κάθε έτος. Άρα στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να αποφανθούμε για το πόσο, τι ποσό θα δαπανάτε κάθε χρόνο. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε και αυτό έγινε και σε ό,τι αφορά το Task Force για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Το πρώτο έτος ήταν μάλλον αργή η εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια επιταχύνθηκε και αυξήθηκε. Άρα, φανταζόμαστε ότι θα ξεκινήσουμε με ένα αρκετά χαμηλό ποσό, το οποίο και θα αυξηθεί σε ό,τι αφορά τη χρήση του τα επόμενα χρόνια κατά τη διάρκεια της τετραετούς περίοδου. Τώρα, να δούμε δύο πράγματα για τον συντονισμό και τον, ε, τη συμπληρωματικότητα. Σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή τώρα, ξέρουμε ότι η τεχνική αρρωγή λαμβάνει η χώρα και σε άλλα πλαίσια. τεχνική αρρωγή σε διάφορα διάφορα ταμεία. Και γίνεται αυτό φυσικά με, μέσω άλλων τμήματων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω άλλων κρατών μελών. Αυτό λοιπόν που τονίζουμε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος είναι ότι δεν θέλουμε αλληλεπικαλύψεις, δεν θέλουμε ε, αλληλεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια που παρέχεται. Θέλουμε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που είναι στη διάθεσή μας προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, γίνεται ένας συντονισμός και ακολουθούμε την προσέγγιση της φιλογραμματικότητας. Τι σημαίνει αυτό. Ανάλογα με τα αιτήματα που λαμβάνουμε, η πρώτη αντίδραση στο κάθε αίτημα είναι να ελέγξουμε και στις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα κρατημέλη κατά πόσον ήδη έχει χορηγηθεί τεχνική αρρωγή στους τομεί αυτούς, προκειμένου, όπως είπα, για να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν Το σημείο λοιπόν που τονίζουμε εδώ είναι ότι θέλουμε να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ένα άλλο δε στοιχείο της πρότασής μας. Και αυτό γιατί οι πόροι που που χρησιμοποιούνται είναι μάλλον περιορισμένοι σε σύγκριση με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή δηλαδή χρηματοδότηση. Άρα, με την τεχνική βοήθεια, την τεχνική αρρωγή που παρέχουμε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε συνεργασίες, συνεργίες, σαν να πούμε καλύπτουμε τα κενά όπου υπάρχουν να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχουν άλλοι τομείς όπου η τεχνική αρρωγή θα μπορούσε να ωφελήσει πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά και τις διάφορες μορφές συνέργειας που μπορεί να διαμορφωθούν. Και προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, έχουμε εφαρμόσει και υλοποιούμε ένα μηχανισμό συντονισμού, έναν εσωτερικό μηχανισμό συντονισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει σαφήνεια ότι είναι ξεκάθαρο το τι έχουμε ήδη πετύχει, τι έχουμε δώσει ήδη και πού εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Επίσης, ο συντονισμός έχει να κάνει και με το τι παρέχεται εξωτερικά στα κράτη-μέλη ως προς την τεχνική αρρωγή από διεθνείς οργανισμούς, ώστε ούτε εκεί να υπάρχουν επικαλύψεις αν έχουν λάβει δηλαδή τα κράτη-μέλη αρρωγή από διεθνεί οργανισμού. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε στο πλαίσιο της ε, υλοποίησης της ε, τεχνικής αρρωγής. Η τεχνική αρρωγή δεν παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους. Η ευθύνη για τη χρήση της τεχνικής αραγής προκειμένου να υποβοηθηθούν οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη είναι στα χέρια του κράτους μέλους. Το γεγονός δε ότι παρέχεται τεχνική αρρωγή δεν σημαίνει ότι υπάρχει παρέμβαση και δεν τηρείται η επικουρικότητα του κράτους μέλους σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων αυτό που ελπίζουμε όλους ιδιαιτέρως, και αυτό πραγματικά αποτελεί σημείο κλειδί είναι το εξή. Η τεχνική ρογή που παρέχουμε να μπορεί να αξιοποιείται, να είναι ωφέλιμη. Να μην βρεθούμε σε κατάσταση όπου θα καταλήξουμε να έχουμε απλά εκθέσεις οι οποίες θα μπαίνουν σε ένα και τελείωσε. Αυτό που μας απασχολεί λοιπόν όλος ιδιαίτερος είναι να παρέχουμε τεχνική αρρωγή η οποία πρακτικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη για να υποβοηθηθούν. Και στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία μεταρρύθμισης εξακολουθεί να μένει αποκλειστικά και μόνο στα χέρια του κράτους μέλους. Η πρόταση τώρα αυτή μας επιτρέπει να καταρτήσουμε και δείκτες και να κάνουμε και μια αξιολόγηση. Όταν χορηγείται τεχνική αρρωγή σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, ασφαλώς και παρακολουθούμε την τεχνική αρρωγή που παρέχεται για να εξασφαλίσουμε ότι επιτυχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Υπάρχει λοιπόν μια διαρκής διαδικασία παρακολούθησης σε σχέση με τα όσα είχαν συμφωνηθεί για τα για τους στόχους και κατά πόσον έχουν πραγματικά επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί. Άρα, οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα συμπεριλαμβάνονται σε κάποιους ποιοτικού δείκτες που προβλέπονται για το πρόγραμμα. Άρα, οι ενέργειες περιλαμβάνουν παροχή εμπειρογνωμοσύνης, ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη, όλους αυτούς τους στόχους τους που έχουν τεθεί στη, στα πλαίσια της ε, αρρωγής. Οι ποιοτικοί δείκτες έχουν να κάνουν με το feedback, στατικό και δυναμικό από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων για την, ε, τον αντίκτυπο της τεχνικής αρρωγής. Τι θέλω να τονίσω εδώ. Ότι δεν θα δώσουμε απλά τεχνική αρρωγή και, και τελειώνει η υπόθεση. Όχι, μας απασχολεί και η αξιολόγηση, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να είναι ικανοποιημένοι και ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς με την τεχνική αρρωγή που λαμβάνουν. Και επίση θα θέλαμε να δούμε πώς αξιοποιείται, πώς χρησιμοποιείται στην πράξη αυτή η τεχνική αρρωγή. Το τμήμα της αξιολόγησης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό της όλης διαδικασίας. Ως προς την αξιολόγηση, πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα Έχουμε προβλέψει μια διάμεσα αξιολόγηση μέχρι το τέλη του 2019 και τέλος, στο τέλος της τετραετούς περίοδου προφανώς προβλέπεται και μια εξπόστα αξιολόγηση το 2021 δηλαδή. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε ό,τι αφορά την πρόταση. Στην παρούσα φάση έχει βελτιωθεί η έχει εγκριθεί μάλλον η πρόταση από την Κορεπέρ στις 28 Μαΐου συγκεκριμένα μετά από μια σειρά τεχνικών συναντήσεων με, του, με την ομάδα εργασία των δημοσιονομικών συμβούλων και με κάποιες ε, τροπολογίες και προσαρμογές της αρχικής ε, πρότασης. Επίσης, η, η ESC χορήγησε σχετική γνωμοδότηση στις 3 Μαρτίου και η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότηση στις 8 Απριλίου, το τελευταίο σημείο. Και εδώ προφανώς η πρόταση βρίσκεται στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλέον, στην Επιτροπή Ρέτζη, η οποία και είναι αρμόδια και συναρμόδιες είναι και άλλες επιτροπές. Προγραμματίζονται περαιτέρω συναντήσεις και συνεδριάσεις με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές τους ερχόμενους ε, μήνες και κάτι που θα ήθελα να θα αναφέρω σε σχέση με την πρόταση. Η χρηματοδότηση θέλουμε να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Πρώτου του 2017, προκειμένου να υπάρχει αυτή η τετραετής περίοδος για την υλοποίηση του προγράμματος. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια τεχνική συζήτηση επί της πρότασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία και την ημερομηνία αυτή. Και ως εκ τούτου, με χαρά μου είμαι εδώ σήμερα και θα χαρώ να απαντήσω ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Μαζί με τους συναδέλφους εδώ, εξ αριστερών. Έχουμε μαζί μας ε, έναν συνάδελφο ειδικό για θέματα νομικά και την συνάδελφο η οποία είναι ειδική σε θέματα προπολογισμού και χρηματοδότηση. Ευχαρίστω λοιπόν να απαντήσουμε σε όποια ερώτηση ενδεχομένω έχετε. Ευχαριστούμε κυρία Μακάρτη. Ξεκινάμε από το μηδέν. Έχω στον κατάλογο μου δύο ομιλητές, αλλά θέλω να επανέλθω ε, στους προηγούμενους αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Κοιτάξτε, μπορείτε αν θέλετε ε, να κάνετε μια ερώτηση κύριε Σόγκο και να έχετε αμέσως την απάντηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Σόγκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω βασικά δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει μια σε δυσκολία στις ε, εκθέσεις αυτές, ε, μάκρο και μικροοικονομική προσέγγιση και στις δύο προτάσεις είναι ακριβώς η ίδια και εσείς ε, πώς προτίθεστε να επιλύσετε αυτό το θέμα, κυρίως όσον αφορά στη διάθεση των κονδυλίων και δεύτερον πώς θα μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι θα επωφεληθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση από αυτή τη στήριξη και όχι μόνο οι κεντρικές κυβερνήσεις. και κυρία Χάρκινγκ, δεν ξέρω, θέλετε τώρα να ρωτήσετε, όχι θα ρωτήσω στο τέλος, ε, θα πρέπει να φύγω για πέντε λεπτά και στο τέλος της συζήτησης ε, θα επανέλθω. Στον κύριο, ο κύριος Γκουτιέρες Πιέτρο, έχει το Ευχαριστώ και θερμά, θερμά ευχαριστώ προς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες ε, για το ταμείο αυτό και την ουσία, την, το νόημά του. Ε, βέβαια η παροχή τεχνικής συνδρομής ε, δεν είναι αφ' κάτι κακό, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ. Έχω κάποιες ε, αμφιβολίες τις υποβάλλουμε κιόλα, γιατί από τη στιγμή που αφιερώνονται κονδύλια τεχνικής αρρωγής ε, δεδομένου του δημοσιονομικού πλαισίου, είχαμε πρόβλημα σε πολλές περιφερειακές και εθνικές αρχές. Δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία, τα καινούρια κονδύλια. Και μάλιστα όσο προχωρεί το πολιτικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τόσο πιο δύσκολο είναι για τα περιφερειακά όργανα και τα εθνικά να δικαιολογήσουν αυτά τα ταμεία. Τώρα, έχουμε πιο περίπλοκα προγράμματα που παρέχουν συνδρομή και ταμεία, όπως το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν είμαι βέβαιος ότι το νέο Ταμείο Στήριξης ε, είναι κατάλληλο, γιατί είναι τόσο περίπλοκες οι αλλαγές και από την προηγούμενη και από την τωρινή κοινοβουλευτική θητεία τώρα το να διευρύνουμε τη συνδρομή και προς άλλες χώρες με τόσο σημαντικές διαφορές δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Από αυτό που τεχνική άποψη μια επιφύλαξη τεχνικής φύσεως, δηλαδή να, να αφαιρέσουμε κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να χορηγήσουμε πολιτική συνδρομή, γιατί περί πολιτικής συνδρομής πρόκειται γιατί είναι πολιτικά αυτά τα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Έχω λοιπόν πέραν των τεχνικών επιφυλάξεων και κάποιες πολιτικές επιφυλάξεις. Όταν μιλούμε για κονδύλια που παρέχουν αρρωγή στα κράτη-μέλη για την διεξαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ερχόμαστε σε προηγούμενες ε, εποχέ που μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μερικέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις είχαν αντικυκλικά αποτελέσματα και ουσιαστικά βάθαιναν την ύφεση. Και κάποιε χώρε χρειάστηκαν κονδύλια για να αντισταθμίσουν αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να μην επιβαρύνουν περαιτέρω του πολίτε. Οπότε αυτό το Ταμείο τεχνική συνδρομή χρειαζόταν, αλλά με τη μορφή περισσότερο οικονομική αρρωγή, ε, κοινωνική αρρωγή. και τα 142 και κάτι εκατομμύρια δεν αρκούν για κάτι τέτοιο. Πέραν του πολιτικού προβλήματος υπάρχει και ένα πρόβλημα κοινωνικό. Γιατί πολλοί συμπολίτε μας, κυρίως από την Νότια Ευρώπη, σε χώρες που χρειάστηκε να κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ε, πώς αντιλαμβάνονται την τεχνική σύνδρομη για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Την αντιλαμβάνονται ως περικοπές. Περιστολές δαπανών και περικοπές ε, των κοινωνικών ε, παροχών. Τώρα, αν ε, δημιουργήσουμε ένα ταμείο που θα δίνει συμβουλές στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, θα θορυβήσει ακόμη περισσότερο του συμπολίτε μας που ήδη φοβούνται αυτή τη τεχνική συνδρομή γιατί την εκλαμβάνουν ως περικοπή του κράτους πρόνοιας. Και ο σοσιαλιστής και εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες. συμφωνώ ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, να εξυγχρονίζουν την οικονομία και να αντισταθμίζουν τις ε, κοινωνικές ε, και οικονομικές αρνητικές συνέπειες της κρίσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευημερία. Αλλά οι πολίτες, βλέποντας τα στοιχεία της Eurostat, δεν σχηματίζουν την εντύπωση ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα έχουν αυτή τη διάσταση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της διασφάλισης της κοινωνικής προστασίας και της ε, κοινωνικής ευημερίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα προσκρούσουμε σε πολλές αντιδράσεις για αυτό το νέο ταμείο. Οπότε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ναι, θα πρέπει να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα συντονισμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά θα πρέπει να δούμε τους στόχους, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε το ευρωπαϊκό εξάμεινο όχι μόνο για θέματα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά για να κάνουμε ένα copy-paste των ε, δράσεων των κρατών μελών παρά τις αλλαγές που έχουμε στο παραγωγικό μας μοντέλο, στις εργασιακές μας σχέσεις, στις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα, αν αυτό το νέο ταμείο, αν αυτή η τεχνική συνδρομή θα χρησιμοποιηθεί μόνο να γίνει ένα copy-paste ε, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κεκτημένα, τα συνδικαλιστικά, κοινωνικά και άλλα, δεν θα μας βρει σύμφωνος μια τέτοια πρόταση. Αν απλώς θέλετε να προσαρμόσετε την πραγματικότητα σε κοινούς στόχους και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στις χώρες τα τελευταία χρόνια με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουν γίνει, ε, επί Επιτροπής Μπαρόσο, και οι εργασιακές και οι ταξιδοτικές μεταρρυθμίσεις είχαν αποτέλεσμα εξίσου. Ίδιο ε, συντάξιμο, ε, ηλικία συντάξιμη και άλλα θέματα φορολογικά ουσιαστικά εξομοίωσαν την κατάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου, ενώ είχαμε χώρες με τελείως διαφορετική δημογραφική, εργασιακή, κοινωνική κατάσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική συνδρομή για να εφαρμόσουμε το ίδιο κουστούμι σε όλους ε, και μια ενιαία αντιμετώπιση σε όλους. Δεν νοείται τέτοια ενιαία αντιμετώπιση με τόσο μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε ούτε συμφωνώ να αφαιρούμε κονδύλια από το κοινωνικό ταμείο για να πρικοδοτήσουμε αυτό το ταμείο και να δίνουμε τεχνική συνδρομή ε, για την Ενεργειακή Ένωση ή για άλλα θέματα που δεν έχουν σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα πρώτα να ορίσουμε τους τεχνικούς ε, στόχους σε επίπεδο πολιτικό. Και παραλαμβάνω να μην κάνουμε ένα απλό, ένα απλό copy-paste ε, συστάσεων για χώρες που έχουν τελείως διαφορετικά και εκτιμένα διαφορετική παράδοση, ιστορία και επιδόσεις ε, και να εφαρμόσουμε τις ίδιες συστάσεις για όλους. Αυτό θα αυξήσει το σκεπτικισμό των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στις ενέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Ε, υπάρχει ακόμα μία ερώτηση, αλλά δεν ξέρω. Μήπως θέλετε να αρχίσετε ήδη να απαντάτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Για να φτάσουμε στη χρηματοδότηση, το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας ευθύς εξ αρχής είναι το εξή. Σε αυτή την ε, ζωφερή οικονομική περίοδο, τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία όρεξη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση. Άρα ε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να επιτύχουμε νέα χρηματοδότηση. Και έτσι ε, το ερώτημα που βάζουμε στον εαυτό μας είναι από πού πρέπει να προέρθει αυτή η χρηματοδότηση. Ε, καταλήξαμε στο να δούμε λιγάκι τα περιθώρια της υπάρχουσας χρηματοδότησης. Εξετάσαμε τους διάφορους τομείς για να δούμε ποια είναι τα περιθώρια. Ε, εξετάσαμε κάθε τομέα μεμονωμένα και κάναμε και μία ανάλυση. Αυτό το έκαναν οι δικοί μας για τα δημοσιονομικά. Εξέτασαν λοιπόν τη χρήση των κονδυλίων ε, των διαφόρων τομέων σε σχέση με τα ανώτατα όρια που προβλεπόντουσαν. Και λήφθη επίσης υπόψη η αύξηση της χρηματοδότησης ε, για διάφορους τομείς. Έχουν αυξηθεί τα ανώτατα όρια για να ληφθούν υπόψη και επιπρόσθετες απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της αξιολόγησης ήταν ότι ε, επί τη βάση της ε, παλαιότερης χρήσης κονδυλίων και επί τη βάση ε, του να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετες ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς, πράγματι στο 1β υπάρχει ένα περιθώριο, από εκεί μπορούμε να πάμε κάποια κονδύλια να πάρουμε κονδύλια για να ε, χρηματοδοτήσουμε τα δικά μας τα προγράμματα. Κάναμε τη σχετική ανάλυση για τις ε, παλαιότερες ε, τάσεις και έχοντας κατά νου και την προβλεπόμενη αύξηση αναγκών των κρατών μελών στην τρέχουσα περίοδο. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι τα απαραίτητα ποσά μπορούσαν να ε, αφαιρετούν από αυτό τον τομέα που σας είπα χωρίς να συρρυκνώσουμε και να συμπιέσουμε ε, ανάγκες σε συγκεκριμένες τομείς. Όλα αυτά έγιναν επί τη βάση μιας υγιούς μελέτης. Το άλλο το οποίο θέλω επίσης να υπογραμμίσω είναι ότι πράγματι τα κονδύλια εκταμιεύονται ε, σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα λοιπόν εμείς περιλαμβάνουμε και άλλους τομείς ε, κυρίως όσον αφορά την τεχνική αρρωγή, αλλά αν δει κανείς τους τομείς που καλύπτονται ε, στο ε, EFSF και σε άλλα ταμεία, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει επικάλυψη τομέων. Έτσι λοιπόν, ο μόνος τομέας ή οι μόνοι τομείς για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε και που να αφορούν στη δυνατότητα εκταμίευσης τεχνικής αρρωγής είναι τομείς όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας και επίσης ε, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι όσον αφορά τη χρήση της ε, τεχνικής αρρωγής, κονδύλια επίσης μπορούν να προβλεφθούν για τεχνική αρρωγή ε, για θέματα που έχουν σχέση με τη μετανάστευση. Και αυτή τη στιγμή αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα σε αυτό ε, για το οποίο θα χρησιμοποιούνταν αρχικά τα κονδύλια και στο τι τελικά χρησιμοποιούνται. Εγώ δεν ε, βλέπω να υπάρχει ε, κάποια συγκεκριμένη σύγκρουση σε σχέση με, τους, με την προβλεπόμενη χρήση των κονδυλίων. Τώρα όσον αφορά τα ωφέλη, τα τοπικά ωφέλη, είναι αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται να λειτουργούμε είναι ο εξής. Λόγω της φύσης της ε, δουλειάς μας, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρχές ε, τα κράτη-μέλη το αίτημα τεχνικής αρρωγής μπορεί να καλύπτει πολλούς τομείς, ε, παραδείγματος χάρη ε, μπορεί να καλύπτει και τοπικά θέματα. Για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό. Ένας από τους βασικούς τομείς ε, παρέμβασης ε, για τεχνική αρρωγή κατά το παρελθόν ήταν η δημόσια διοίκηση. Το να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ε, δημόσιας διοίκησης, αυτό είναι ένα σημαντικό σκέλος της τεχνικής αρρωγής ε, που χορηγήθηκε κατά το παρελθόν. Και βεβαίως και αυτό δεν αφορά μόνο στην δημόσια διοίκηση σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και στη δημόσια διοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά στους ε, τομείς για τους οποίους μπορεί να προσφερθεί τεχνική αρρωγή. Εδώ μιλάμε για όλες τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει μία χώρα είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εμείς ε, θεωρούμε ότι αν και το διοικητικό σκέλος αφορά την κεντρική διοίκηση, παρόλα αυτά ε, δεν έχει επιπτώσεις για το πού ακριβώς προσφέρεται η τεχνική αρρωγή. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει συντονισμό σε κεντρικό επίπεδο, είτε διαπραγματευόμεθα διμερός, είτε διαπραγματευόμεθα με μια συγκεκριμένη αρχή, φορέα, που είναι αρμόδιος ε, για αυτή τη συγκεκριμένη αρρωγή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά την απάντηση στην ερώτηση για τα τοπικά και περιφερειακά ωφέλη. Όσον αφορά τώρα στο θέμα της ουσίας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι ο εξής. Έχουμε ένα συγκεκριμένο επιμερισμό εργασιών για το πώς ακριβώς λειτουργούμε. Δηλαδή, Έχουμε τις ε, συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κράτους μέλους και αυτή είναι μια συμφωνία που δεν είναι υπό την δική μας την αρμοδιότητα. Βεβαίως, ε, τα κράτη-μέλη ε, καθορίζουν μόνα τους τις προτεραιότητες τους. Συμφωνούν ή αποφασίζουν για τις διατροτικές τους μεταρρυθμίσεις ε, και από τη στιγμή που το κάνουν ζητούν από μας βοήθεια για την ε, ε, εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αν το κράτος μέλος θέλει βοήθεια, το ζητάει. Αν όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς, δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, θέλω να πω, δεν μπαίνουμε σε πολιτικό, πολιτική διαμάχη. Εμείς δουλεύουμε καθαρά σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας. Και κάτι άλλο που θέλω να σκεφτείτε είναι το εξής. Ε, πρόκειται για τη φύση της ε, τεχνικής αρρωγής. Για μας δεν είναι μια τεχνική αρρωγή που ταιριάζει για όλους. Δεν υπάρχει μαγική απάντηση για το καλύτερο είδος τεχνικής αρρωγής. Αυτό που αποδίδει σε ένα κράτο μέλος μπορεί να μην αποδώσει σε άλλο. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα τεχνική αρρωγής για μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η πρώτη μας απάντηση είναι να κάτσουμε με το εν λόγω κράτος μέλος, τις αρμόδιες αρχές, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς επιθυμεί ε, να επιτύχει το κράτος μέλος. Μπορεί ε, να έχουν κάποια ιδέα για το σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, μπορεί και όχι. Ίσως να υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις για τη μεταρρυθμίση και σε τελική ανάλυση το κράτο μέλο είναι εκείνο που λαμβάνει την τελική απόφαση. Τίποτα δεν επιβάλλεται στο κράτο μέλο ως προς το σχεδιασμό. Επίσης, όσον αφορά τη μορφή της τεχνικής αρρωγή και αυτό ε, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους. Παραδείγματο χάρη, για να έχετε έτσι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένα κράτος μέλος ε, ήθελε να ανασχεδιάσει το σύστημα της ε, κοινωνικής ασφάλισης και να εισάγει ε, εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα έτσι ώστε στη χώρα αυτή να προσφέρεται ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αφού ετέθη το αίτημα αυτό, εμείς ρωτήσαμε πώς θέλετε να ορίσετε τις ε, παραμέτρους αυτού του μέτρου. Εσείς θα το κάνετε, το, εσείς θα ορίσετε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και αφού γίνεται αυτό, μετά εμείς εξετάζουμε ε, διαφόρους ε, που μπορούν να βοηθήσουν το κράτος μέλος. Δεν λέμε ότι να απευθυνθείς ε, εδώ ή εκεί παραπέρα, αλλά δίνουμε την αναλλακτική λύση στο κράτος μέλος για το που πρέπει να στραφούν έτσι ώστε να εφαρμόσουν αυτή τη συγκεκριμένη διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Άρα δηλαδή σας λέω είναι καθαρά διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Και η εμπειρία που έχω κάνει είναι ότι όταν μιλάμε για βέλτιστες πρακτικές, ε, δεν είναι απαραίτητο οι βέλτιστες πρακτικές ενός κράτους μέλους να είναι ίδιες και σε ένα άλλο. Αυτό που λειτουργεί σε ένα κράτος μέλος, ε, αν δει κανεί τις συγκεκριμένες παραμέτρους και τις ε, συνθήκες που επικρατούν, δεν ισχύει απαραίτητα και για άλλο κράτος μέλος. Δεν είναι δηλαδή ένα μοντέλο που μπορεί να ταιριάξει και σε άλλο κράτος μέλος. Άρα δηλαδή εσείς έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τις ε, παραμέτρους για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, εμείς ε, δεν επιμένουμε στο να εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά βρίσκονται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας. Ε, τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος Πυρίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση κανονισμού ε, μας δίνει πολύ τροφή για σκέψη και θεωρώ ότι χρήζει πολύ μεγαλύτερης προσοχής και από την Επιτροπή Απασχόλησης. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε μια έξοδο των βουλευτών από την Επιτροπή με αποτέλεσμα να μείνουμε τρεις και ο κούκος στη συζήτηση. Η πρόταση έγινε μια σειρά θεμάτων και ερώτημάτων. Οι εκτενείς και αδελεχείς απαντήσεις και διευκρινήσεις που μας έδωσε η κυρία Μαγκρέγκορ και στην αρχική παρουσίαση και στις απαντήσεις τροφοδοτεί μια νέα πληθώρα ερωτήσεων. Θα ήθελα καταρχήν να διαπιστώσω κάτι που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η χρήση των κονδυλίων περνά από ένα πλαίσιο σε άλλο. Και τα κονδύλια αυτά στις συνθήκες περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η νομική βάση για την πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, είναι το άρθρο 175, παράγραφος 3 Πολύ περίεργη η διατύπωση του κειμένου. Γιατί παίρνουν το τίτλο και των μέσων, αναφέρει ως σκοπό την προώθηση τη συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και την υστέρηση των μειονεκτικών περιοχών, των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Και στην τρίτη παράγραφο του 175 άρθρου αναφέρεται ότι αν χρειαστούν ε, συγκεκριμένες δράσεις εκτός των κονδυλίων και των ταμείων που προβλέπονται στον τίτλο αυτό και υπό την επιφύλαξη των μέτρων που εγκρίνονται στα πλαίσια άλλων πολιτικών, τέτοιες δράσεις ε, ίσως ε, υιοθετηθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, συμπληρωματικέ δράσει πέραν αυτών που προβλέπονται στα ταμεία και κονδύλια, αλλά και πάντα στο πλαίσιο τη συνοχή και όχι άσχετα με τη συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε διαφορετική ερμηνεία αυτού του άρθρου και λέει όχι μόνο θα έχουμε συμπληρωματικέ δράσει εκτό των ταμείων αυτών, αλλά και θα αφαιρέσουμε από το ταμείο ε, το κοινωνικό θα τα διαθροτικά, κάποια κονδύλια και θα τα βάλουμε σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ δημιουργική και ευρηματική αφενός, αλλά και ιδιαίτερα παράλογη και αλλοπρόσαλη ερμηνεία του άρθρου για τη δημιουργία αυτού του νέου προγράμματος. Και μάλιστα φαίνεται ότι δηλείται έμπνευση για το πρόγραμμα αυτό από τις εμπειρίες που αποκομίσατε από τα προγράμματα της ε, Ελλάδας και της Κύπρου. Και αυτή η πηγή έμπνευσή σας μου φαίνεται κάπως περίεργη. Γιατί τα προγράμματα που εφαρμόζουν ακόμη δύο χώρες, ειδικά η Ελλάδα, έγιναν υπό ε, έκτακτες περιστάσεις, ε, ιδιαίτερων αντικσότητων και δυσκολιών. Και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πάνω κάτω υπαγορεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε μεγάλο βαθμό το έργο των, της γνωστής Τρόικας. Και δεν ήταν και πολύ δημοφιλής για να μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι μόνο στο λαό των χωρών αυτών, αλλά και γενικώ στην Ευρώπη δεν ήταν καθόλου δημοφιλή αυτά τα μέτρα και αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί θεωρήθηκε ότι δεν βοηθάνε στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Και όχι μόνο δεν βοηθούν, διόρθωση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά οδηγούν οικονο... τις οικονομικές πολιτικές σε τελείω λάθος κατεύθυνση. Χθε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη είχαμε συζήτηση επ' ευκαιρία μιας ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τη δημιουργία οικονομική ανάπτυξη ε, στα πλαίσια του παραγράφου, της παραγράφου 16 του CPR. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η συνοχή και η σύγκληση διακόπησαν μετά την κρίση του 2008 και του 2009 και αντί να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση έχουμε όλο και μεγαλύτερη απόκληση. Οπότε σίγουρα έχουμε σοβαρές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και βασικότερη είναι να επιστρέψουμε στην πορεία της συνοχή. Ε, και Εξετάζοντας την τεχνική συνδρομή που προσφέρεται στους διάφορους τομείς, ε, στόχος έπρεπε να είναι η πρόθεση της συνοχής και κανένας άλλος σκοπός από την πληθώρα στόχων προσπαθείτε να υλοποιήσετε μέσω αυτής της τεχνικής συνδρομής. Έχουμε τις ειδικές τέσσερα χώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στα πλαίσια αυτών ίσως χρειαστεί κάποια τεχνική συνδρομή. Αλλά το να συγχαίουμε τα δύο πράγματα είναι τελείως απαράδεκτο. Και είναι περίεργο που βάζετε χέρι σε ταμεία, ακόμη και σε, στο ταμείο για τους απόρους, το κοινωνικό ταμείο. Πριν από δύο μέρες μας επισκέφθηκε στην Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και η Επίτροπος Στάισεν και μας είπαν ότι ήδη υπάρχει μεγάλη ανάγκη και τα ταμεία είναι πολύ, ε, σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν υπάρχουν επιπλέον κονδύλια. Και προτάθηκε αύξηση των ανώτατων ορίων. Αλλά υπάρχει απροθυμία γι' αυτό και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και την υπαρξιακή κρίση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι οι προτάσεις σας θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερα επιχειρήματα για την ε, ενίσχυση της ε, πλευράς της αποχώρησης ε, του, Ευρωπα... του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ρίξουν νερό στο μήλο αυτών που ζητούν τον Brexit. από ποιες, ε, από ποια κονδύλια της συνοχής θα αφαιρεθούν για το νέο πρόγραμμα από τους 15 ε, συν είμαι κατά της εξαγωγής κονδυλίων συνοχής για την χρηματοδότηση του προγράμματος ε, τεχνικής συνδρομής. Και μάλιστα ήμασταν κατά και της αφαίρεση κονδυλίων από το συνδέοντα στην Ευρώπη για να τροφοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το είχαμε πει κατηγορηματικά και ζητήσαμε την επαναφορά των κονδυλίων στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Και όχι, αντί να εισακουστεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ακόμα μεγαλύτερη αφαίρεση κονδυλίων. Προσοχή λοιπόν σε τέτοιο είδου προτάσει. Εγώ θα πρότεινα να προγραμματίσουμε και νέα συζήτηση για το θέμα αυτό και θα έλεγα η Γραμματεία να καλέσει τους Ευρωβουλευτές να υποβάλουν ερωτήσεις και να έχουμε και δεύτερη συζήτηση με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όποιο επίπεδο κρίνουν ότι είναι απαραίτητο μετά την λήψη όμως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των γραπτών της απαντήσεων. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, αυτή η πρόταση ακούγεται καλή. Θα το συζητήσουμε ενδεχομένω στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα το συζητήσουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουμε άλλη μία που προβλέπετε πριν από τις θερινές διακοπές. Δεν είχαμε ως τώρα το χρόνο και την ενέργεια να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Πριν από τις ε, θερινές Και όπως βλέπετε, είναι έντονες οι αντιδράσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση. η οποία θα συνάδει και με το πολιτικά υπεύθυνο σκέλο τη επιτροπή. Δεν σα έκανε ερωτήσει ο κ. Πυρίνσκι, αλλά φυσικά μπορείτε να πάρετε το λόγο για να συνοψίσετε και να μα παρουσιάσετε τι δικέ σα θέσει. Ναι, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια ζητήματα, αν με επιτρέπετε. Και οι εμπειρογνώμονε, μάλιστα, θα ήθελα να πάρουν το λόγο για να διευκρινίσουν ενδεχόμενε παρανοήσει. Να ξεκινήσουμε από τις νομικές υποθέσεις, τα νομικά ερωτήματα. Ο γενικός στόχος ε, της πρότασης αναφέρει ως γενικό στόχο της αρρωγής την υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη προκειμένου οι εθνικές αρχές ε, της ε, χώρας πέρα από την κεντρική κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, δηλαδή να υπάρξει μεταρρύθμιση της διοίκησης του οικονομικού και κοινωνικού τομέα. σε ό,τι αφορά και τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει και την στοχευμένη χρήση των κοινωτικών πόρων. Οι κοινωτικοί πόροι που αναφέρονται στο πλαίσιο του CSSP ασφαλώς είναι το ΕΣΥΦ, τα τροφωτικά ταμεία, αλλά και ταμεία τα οποία δεν είναι διαφορετικά ταμεία. αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν όπως ε, τα ταμεία, όπως για παράδειγμα τα ταμεία για τη μετανάστευση, για τους πλέον ενδεείς, όπου δεν αφαιρούμε χρήματα πόρους από τα ταμεία αυτά, αλλά ως γενικό στόχο του προγράμματος παρέχουμε την ευκαιρία να βοηθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κράτη-μέλη. Και αναφέρομαι στο γενικότερο στόχο, τον απότερο στόχο, γιατί προφανώ η συνοχή είναι πολύ σημαντικό σκέλο. Γιατί έτσι, με τον γενικότερο στόχο του SSP, συμβάλλουμε στην επίτευξη του γενικότερου στόχου της Συνθήκης Λισαβόνας που ορίζεται στο άρθρο 174 και είναι η συνοχή. Αυτός λοιπόν είναι ο απότερος στόχος του CSSP. Και μιας και θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο της συνοχής που ορίζεται στο 174 άρθρο, θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό όπου θα μπορούσαμε να δράσουμε πέρα από τα τα ταμεία που ρυθμίζονται από το άρθρο 177 της συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου ακριβώς να πετύχουμε τον στόχο της Λισαβόνας για την Λισαβόνα. 175 άρθρο, παραγραφός 3, όπως αναφέρατε αξιότιμη κύριε Βουλευτά Πρίνσκι. Το 175 λοιπόν αφορά τα κράτη-μέλη και το ρόλο που παίζουν για την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και προαπαιτεί το άρθρο αυτό και προδιαγράφει την κατάρτιση των σχετικών οικονομικών πολιτικών και τον έλεγχο των πολιτικών αυτών για να επιτευχθεί ο στόχος της συνοχής. Σε περίπτωση που η, η Ένωση θεωρεί ότι ενδεχομένω υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να λάβουν χώρα πέρα από τα ταμεία αυτά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μπορεί να γίνει πρόταση κανονικής νομοθετικής ε, διαδικασίας για την επιτεύξη των στόχων αυτών του άρθρου 175. Ακριβώς αυτό κάνουμε με την πρόταση αυτή. Προφανώς ε, αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο στόχο της ε, πολιτικής συνοχής και των όσων θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με το CSISP το οποίο συνάδει με το γενικότερο στόχο. Υπάρχει και άλλη μια νομική βάση, το άρθρο 197. Ο λόγος που υπάρχει διπλή νομική βάση στην πρότασή μας είναι αυτός που ανέφερε και η κυρία Μακάρθη. Ο λόγος είναι ότι δεν βοηθάμε μόνο τα κρατημέλη δεν περιοριζόμαστε στο στόχο της συνοχής μόνο, γιατί θέλουμε να ανταποκριθούμε στο αιτήμα των κρατών μελών για να παρέχουμε βοήθεια που δεν καλύπτεται από τα υπόλοιπα άρθρα. Και γι' αυτό λοιπόν το άρθρο 197 καλύπτει την διοικητική συνεργασία για τη συνεργασία σε κοινωτικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν βάσει αυτού μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε κράτη-μέλη που, για στόχους που δεν καλύπτονται από τη συνοχή. Για παράδειγμα, για τη μετανάστευση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στη συνοχή, αλλά θέλουμε να παρέχουμε αρρωγή, γιατί είναι τεράστιε οι ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το διοικητικό σκέλος για τη μετανάστευση. Δεν θα μπορούσαμε να την παρέχουμε την αρρωγή αυτή, αν είχαμε περιοριστεί μόνο στη νομική βάση του 175 άρθρου και του 174 ως προγραμματικά στοιχεία. Ε, έπρεπε να υπερβούμε το επίπεδο αυτό και γι' αυτό λοιπόν από νομική άποψη επιλέξαμε τη διπλή νομική βάση και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η αντίδραση για να καλύψουμε ακριβώ του τομεί όπου ενδεχομένω να ανακύψουν ανάγκε από πλευρά των κρατών μελών. Θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσω κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι το CPA καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο, παντελώς καινούριο για τα διαρθρωτικά ταμεία και καθιστά σαφή τη σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση. Διότι όπως αναφέρεται στο κείμενο, αν δεν υπάρχει σε οικονομική διακυβέρνηση που να στηρίζει τα διαρθρωτικά ταμεία, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική χρήση αυτών των κοντιλίων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους των διαρθρωτικών ταμείων. Άρα υπάρχει διασύνδεση και υπάρχει και με το άρθρο 175 παράγραφο 1 όπου αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν την οικονομική τους πολιτική να την εφαρμόζουν με τέτοιο τρόπο που αυτή να συμβάλλει στην πολιτική συνοχή. Και, τα, και η Κομισιόν οφείλει να στηρίζει τα κράτη-μέλη σε αυτή τους την προσπάθεια. Δεύτερον, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε και δεν παίρνουμε χρήματα από τα τους εθνικούς φακέλους όπως λέγονται για την τεχνική αρρωγή είναι μόνο η αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό που προέρχεται από την τεχνική αρρωγή της Κομισιόν για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν τα εθνικά τους προγράμματα ε, και βεβαίως και την αξιολόγηση κτλ. Άρα δηλαδή τα κονδύλια αυτά είναι τόσο μικρά που πραγματικά δεν επηρεάζουν επουδενή την εφαρμογή και το σεβασμό των στόχων των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Χωρίς υγιείς οικονομικές πολιτικές δεν μπορεί κανείς να επιτύχει ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να επιτύχει υγιείς αγορές εργασίας, δεν μπορεί να επιτύχει όλα αυτά για να μειώσει τις ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου να έχει ε, επιτυχή ε, λειτουργία και χρήση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Νομίζω όλα αυτά αποδεικνύουν την χρησιμότητα αυτής της έκθεσης. Έχουμε ένα κράτος μέλος το οποίο μας δίνει χρήματα από τη δική του την τεχνική βοήθεια ε, για να είναι πιο αποτελεσματική βοήθεια και για να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στα κράτη-μέλη. Δίνουν λοιπόν τα δικά τους χρήματα, μα δεν αποδεικνύει αυτό πόσο χρήσιμο είναι να ε, κάνει η Κομισιόν αυτή τη δουλειά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της την τεχνική αρρωγή με τα δικά της τα χρήματα θέλει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Εσείς επίσης επισημάνατε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος κάτω από τελείως ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες και θέλουμε να εμποδίσουμε άλλα να βιώσουν στο μέλλον τέτοιου είδους ακραίες οικονομικές συνθήκες, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε εκ των προτέρων. Και θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρχει ένας γόνιμος προβληματισμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, χαιρετίζουμε, καλωσορίζουμε τους επισκέπτες από το Magdeburg που έρχονται στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά ξέρετε, αργήσατε να έρθετε. Ε, κανονικά αυτή η αίθουσα ε, βρήθη εδώ από ευρωβουλευτές κατάμεστη είναι η αίθουσα υπό συνθήκες, αλλά τώρα τελειώνουμε. Κλείνουμε σιγά σιγά τη συνεδρίασή μας. θα δείτε έτσι, θα πάρετε μια γεύση από το τι συμβαίνει εδώ. Και να δώσω το λόγο για λίγα λεπτά στον κύριο Σόγκορ για να μας πει πώς θα, θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση πρώτα. Αυτή είναι η πρώτη μας ε, συνάντηση, συνεδρίαση. Θα έχουμε και συνεδρίαση με τους συντονιστές, ε, με τους ε, σκιώδης ηγητές, συγγνώμη. Εκεί θα επισέλθουμε στην ουσία και θα εξετάσουμε δελεχέστερα τις αμφιβολίες και τον προβληματισμό της επιφυλάξης. Ωραία. Οπότε εσείς ο εισηγητής θα συναντηθείτε με τους σκιώδεις ηγητές, θα εξετάσετε το θέμα εκτενός και εμβριθός και θα συνεχίσουμε σε επόμενη ευκαιρία τη συζήτηση στους συντονιστές γιατί είναι προφανές ότι θέλουμε να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία και αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ ε, για την προσπάθεια που κάνετε να απαντήσετε σε αυτή την πληθώρα ερωτήσεων. Όπως θα διαπιστώσετε ε, είμαστε μια επιτροπή που ασχολείται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό με τα θέματα αυτά, στρατευμένη και θα επανέλθουμε. Η εξέταση της γνωμοδότησης θα γίνει 31 ε, Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει αργότερα κάποια στιγμή. Η εξέταση των τροπολογιών προβλέπεται για τον Οκτώβριο του 2016. Οπότε έχουμε χρόνο για περισσότερες συζητήσεις, για υποβολή δύσκολων ερωτήσεων και ίσως ε, και πιο σφοδρής ε, συζήτησης. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για την παρουσία σας. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης θα γίνει στις 21 Ιουνίου. Θα έχουμε και εκεί ευκαιρία να προσθέσουμε τα σχόλιά μας πριν τις θερινέ μας διακοπές. Σας ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και τους επισκέπτες μας από το Μαγδεβούργο. Παραλαμβάνω, συνήθως ε, η αίθουσα είναι κατάμεστη με πολλούς ευρωβουλευτές, εκπροσώπους ε, ευρέω φάσματος πολιτικών ομάδων και από τις 28 χώρες μέλη. Μην βλέπετε άδεια τα έδρανα σήμερα. Ε, φανταστείτε την αίθουσα όπως κανονικά είναι, δηλαδή κατάμεστη. Και να σας πω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης ασχολείται με τα ποσοστά ανεργίας, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με τα δικαιώματα των συνδικάτων, με το κοινωνικό θεματολόγιο. Σας διαβεβαιώ ότι είμαστε η πιο αμήλικτη επιτροπή από, τα, από την άποψη αυτή και πιο διεκδικητική. Οπότε θα βρείτε πολλούς ευρωβουλευτές, όπως μπορεί να θέσετε ερωτήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε πάντως και κυρίσω το πέρα της συνεδρίασης.